Ένα σημείο η συζήτηση για την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Κορέας. Καταρχήν οι συντάκτες ε, της ερώτησης θα λάβουν το λόγο. Ο κύριος Κασπάρη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και αξιότιμη κύριε Επίτροπε, η συμφωνία με την Νότια Κορέα είναι έτοιμη. Έχουν μονογραφηθεί τα κείμενα. Πολύ ωραία. Όμως ε, έχουμε την εντύπωση ότι κάποια φορά βλέποντας τις λεπτομέρειες ε, ότι ίσως ε, βιαστήκαμε και δεν έγιναν σωστά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι η προκάτοχό σα ήθελε να κλείσει το θέμα σε κάθε περίπτωση για να έχει τουλάχιστον μια επιτυχία κατά τη θητεία τη. γνωρίζουμε πολλές αναλύσεις που έγιναν σχετικά με τα ωφέλη για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και την οικονομία. Οι θετικέ επιπτώσεις είναι στη φαρμακευτική βιομηχανία, στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες. Όλοι αυτοί οι τομείς και πολλοί άλλοι ακόμη ε, θα ωφεληθούν. Όμως ιδιαίτερα η αυτοκινητοβιομηχανία παραπονείται Έχουμε το πρόβλημα ε, με το, την drawback ε, σχετικά με τα ανταλλακτικά ε, που θα κατασκευάζονται στην Νότια Κορέα και έχουμε και τα προβλήματα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που είναι ανεπίλητα. Πρέπει τους επόμενους μήνες ε, με τους ε, μηχανισμούς ε, και τις ρυθμίσεις των διασφαλίσεων να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Όχι μόνο να τα καταπιαστούμε, αλλά να τα λύσουμε. Νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο μπορούμε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας στη συμφωνία αυτή όταν αντιμετωπιστούν τα και επιληθούν τα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, με προσήκη στο κείμενο. Ε, στο ίντερνετ ε, μπορούμε να δούμε τα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εμείς από κοινού μαζί τους ως ομάδα θα επεξεργαστούμε και μαζί σας θα επεξεργαστούμε μια λύση η οποία δεν θα υπονομεύει τα συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο κύριος Λούκας Ούστα, τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, στην παγκόσμια σκηνή εμφανίζονται νέοι παίκτες. Μερικοί μέχρι τώρα θεωρούνταν αναπτυσσόμενε χώρες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας ε, όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο και τι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μεγάλους ανταγωνιστές τη Ε, εδώ υπάρχουν κάποιε. Ε, ε, λέξεις μαγικές που δεν έχουν μπει μέσα στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμοιβαιότητα, ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκό συμφέρον, ε, καταπολέμηση του ντάμπινγκ και των δασμολογικών ε, εμποδίων. Και σε σχέση με την συμφωνία με την Νότια Κορέα που ε, απασχόλησε ε, δύο επιτρέπους, επιτρόπους και κάποιες εθνικές κυβερνήσεις. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της ε, διμερούς συμφωνίας, ότι το 50% των συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Κορέα αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου εισάγονται πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από την Νότια Κορέα προς ε, εμάς, από ό,τι από την Ευρώπη προς την Νότια Κορέα όταν ορισμένες ε, εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να ε, προωθήσουν τις ε, αγοραπολισίες αυτοκινήτων για να αυξηθεί η κατανάλωση. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας την κλώστο κλωστοϊφαντουργία, συγγνώμη, και, την, και τα ηλεκτρονικά. Ποια είναι τα πλέον για την βιομηχανία μας, την ε, γεωργία μας, ε, τα φαρμακευτικά, ε, όταν είναι ελάχιστα τα πλεονεκτήματα για την αυτοκινοβιχανία ή για την αγορά ηλεκτρονικών. Η υπάρχει, ε, υπάρχουν ε, επιλογές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική της ανάπτυξη. Είδαμε όλοι με ελπίδα τη νέα Ευρώπη που δημιουργήθηκε στην Λισαβόνα. Η νέα όμως αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να μην προωθεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον κόσμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερσούν την Boeing ανέδει της Airbus. Ε, η Αργεντινή προσπαθεί να κοιοποιηθεί την Telecom. Ε, η Νότια Κορέα προσπαθεί να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Κίνα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό Πού κινούνται οι δικές μας μεγάλες επιχειρήσεις και οι χιλιάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειες που απειλείται το μέλλον τους, όχι γιατί παράγουν προϊόντα ε, και αγαθά που δεν είναι υψηλής ποιότητας, αλλά διότι τα δικά τους συμφέροντα δεν προωθούνται. Ε, προχωρήσουμε σε βιαστική επικύρωση αυτής της συμφωνίας, κύριε Επίτροπε. Να θέσουμε σε προσωρινή ισχύ την συμφωνία αυτή, εν αναμονή της επικύρωσης. Είναι απαράδεκτο πριν προσδιοριστούν με σαφήνεια οι σχετικές ε, ε, διαδικασίες και η ρήτρα για την ε, η ρήτρα διασφάλισης πριν αξιολογηθεί η σκοπιμότητα ημί της ε, συμφωνίας αυτής να τεθεί σε ισχύ. Μίχαλ, τώρα δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει νέο κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Η συναπόφαση ε, του ε, Κοινοβουλίου δίνει τη δυνατότητα του επαναδημοκρατισμού των αποφάσεων που θίγουν ως εργαζομένους και καταναλωτές στα κράτη-μέλη τους εργαζομένους. Είναι πολύ σημαντική ευημερία για την Ευρώπη. Οι τάσεις του προστατευτισμού πρέπει να καταπολεμηθούν. Οι συμφωνίες, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όπως αυτή με την Νότια Κορέα μπορεί να φροντίσει για ανάπτυξη και απασχόληση. Βέβαια, ε, ανάλογα με τη συγκεκριμένη συμφωνία βλέπουμε ότι κάποιοι τομείς προωθούνται περισσότερο. Εμείς θέλουμε να δράσουμε εξισορροπητικά. Χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό ε, αξιολόγηση αντίκτυπου. Αυτό πρέπει να το κάνει η Κομισιόν. Όμως, ενώ πολλές φορές και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έχουμε ζητήσει την αξιολόγηση, ε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό άλλωστε διατυπώσαμε και ως ομάδα των φιλελευθέρων αυτή την ε, προφορική ερώτηση. Ε, η σύναψη της συμφωνίας ανοίγει προοπτικές σε πολλούς τομείς, στην γεωργία, στο, ε, για παράδειγμα, όμως προβλήματα υπάρχουν στην υφαντουργία, στην βιομηχανία ηλεκτρονικών και στα αυτοκινήτων. Η συμφωνία με την Κορέα είναι η μόνη με αναπτυγμένη χώρα όπου οι επιστροφές δεν απαγορεύονται. Μπορεί έτσι να υπάρχουν ε, ασύμετρα πλεονεκτήματα κόστους για την βιομηχανία της Νότιας Κορέας. Η Κομισιόν είπε ότι θα ε, εισαγάγει προστατευτική ρήτρα η οποία θα προβλέπει ε, αναστολή κάτω από ορισμένα κριτήρια. Χρειάζεται όμως να ξεκαθαριστεί το θέμα και να μπορεί να εφαρμόζεται και στην πράξη δεν επιτρέπεται ε, να ε, χάνουν την αξία τους οι ρήτρες ε, προστασίας γιατί δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις επειδή φαίνεται να υπάρχουν ασύμετρες ρυθμίσεις και επειδή αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο με μελλοντικέ συμφωνίες με την Ινδία ή την ΑΣΕΑΝ θα πρέπει η προστατευτική ρήτρα να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη ε, και να έχει κεντρική σημασία. Καλούμε μέσα στη συμφωνία. Καλούμε την Κομισιόν, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να ληφθεί γρήγορα η απόφαση και γι' αυτό προσωρινή εφαρμογή ε, τη συμφωνίας δεν μπορεί να γίνει. Από συνομιλίε, ξέρω πόσο δύσκολη είναι μετά η εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό ερωτώ την Κομισιόν. Μπορούμε με την εξωτερική υπηρεσία να έχουμε ισχυρότερο ρόλο στην εμπορική πολιτική. Πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στέρντι έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια των οικονομικών εισχρών για μόνο ε, με την άρση των τελωνιακών και εμπορικών φραγμών μπορούμε να αναζωογονήσουμε την οικονομία μας, ε, να, να προαγάγουμε την ανάπτυξη και να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ για την προηγούμενη συζήτηση. Οι ε, Ευρωπαίοι εξαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοκινήτων, ιατρικών συσκευών είναι ορισμένους από τους τομείς που θα υποφεληθούν τα μάλλα από την άρση των μη δεσμολογικών φραγμών. Χρειάζονται διαδικασίες απλούστευσης ε, στην πιστοποίηση, διαφάνεια και προβλεψιμότητα των τιμών. Όλα αυτά θα ευνοήσουν τον καταναλωτή. Και η νοτοικορεατική αγορά ε, με την ειδίκευση που τη χαρακτηρίζει χρειάζεται ε, γεωργικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρέατα, τυριά, ίνο που προστατεύονται από ενδείξει γεωγραφικής προέλευσης. Ακούσαμε πολλά για το ελεύθερο εμπόριο και την αξία μια τέτοια συμφωνία, χρειάζεται διευκρίνηση σε τομεί αυτή τη συμφωνία, η συμπερίληψη κάποιων <coughs> ρητρών ανάκτηση δασμών, θα πρέπει να διευκρινίσετε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ελεύθερου εμπορίου, θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητα και στο αμοιβαίο συμφέρον. Η πιθανότητα επιβάρυνσης τη Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ασαφής και μας προβληματίζει. Θα, βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, διαβεβαίωσε ότι η, Ευρωπαϊκή, η Νότια Κορέα απελευθερώνει το τελωνιακό καθεστώς και το επίπεδο δασμών που επιδοτούνται από την ανάκτηση δασμών ε, αναθεωρείται. Οπότε θα μειωθούν σταδιακά αυτά τα φαινόμενα της ανάκτησης. Ποια είναι τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκρούσει σε ε, άρνηση για τη ρήτρα διασφάλισης θα προτείνει παράταση της ε, μεταβατικής περίοδου. Θέλουμε πολύ ενδελεχή εξέταση αυτής της ε, ΣΕΣ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Δεχούχτ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ευρωβουλευτέ για, ερωτη... για την προφορική ερώτησή του που επιβεβαιώνει το ζωηρό ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Νότια Κορέα. Αυτή θα είναι η πιο σημαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου για την οποία δίνει επίσημα την συγκατάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, Οπότε χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνεται να διαλευκάνω διάφορε πτυχέ τη συμφωνίας αυτή με την προφορική ερώτηση. Δεν πρόκειται να δώσω διεξοδικέ απαντήσεις σε όλε τι ερωτήσει, αλλά πολύ πιθανό να σα ενημερώσω αργότερα με συμπληρωματικέ ερωτήσει. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δεν είναι η μόνη πρώτη που διαπραγματευόμαστε με χώρε Νοτιοανατολική Ασία. Είναι και η πιο φιλόδοξη και, περιεκτική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από διετή περίπου διαπραγματεύσει, άρχισε να ισχύει από τις 15 Οκτωβρίου του 2009. Στη διαπραγματευτική διαδικασία είχαμε στενές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτήν την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το ψήφισμα για την Νότια Κορέα που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2007 και πολλά από τα θέματα του ψηφίσματος καλύφθηκαν στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Η όλη διαδικασία ε, συνοδεύτηκε από διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και ε, μελέτες επιπτώσεων. Και στα τέλη του Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο την απόφαση για να προχωρήσει στην υπογραφή της ε, ΣΕΣ και την ε, έγκριση της. Στόχος είναι να υπογράψουμε αυτή την συμφωνία ΣΕΣ τον Απρίλιο. Αυτή τη στιγμή μάλιστα ολοκληρώνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάλυση. βέβαια η ΣΕΣ ε, προϋποθέτει την επικύρωση από όλα τα κράτη-μέλη πριν τεθεί επίσημα σε ισχύ. Χρειάζεται λοιπόν και η επικύρωση από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, η διαδικασία αυτή ίσως αποβεί χρονοβόρα και ίσω χρειαστεί για να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ενώσο ε, διαρκεί η διαδικασία επικύρωσης. Αυτό θα, θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο μετά από πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν εφαρμοστεί προσωρινά η ΣΕΣ. Και μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο να λάβουμε υπόψη τι παρατηρήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρί να επιτείνουμε όμω τι καθυστερήσει και να εφαρμόσουμε τη συμφωνία αυτή το συντομότερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τι ρήτρε διασφάλιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση κανονισμού τη στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι επόμενε εβδομάδε και ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να υιοθετήσει αυτό το κανονισμό σύντομα, ώστε η εφαρμογή του να συμπέσει στο μέτρο του δυνατού με την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Τα οικονομικά ωφέλη της ΣΕΣ είναι πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανακουφίσει τους ε, εξαγωγούς ε, βιομηχανικών και γεωργικών ε, προϊόντων και θα εξοικονομήσουν 1,6 δις δασμού το χρόνο μετά την άρση των δεσμών από τις πλευράς της Νότιας Κορέας. Επίσης, οι εξοικονομήσεις θα είναι ακόμη ψηλότερες, γιατί το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Νότιας Κορέας θα αυξηθεί. Με βάση μια μελέτη, η ΣΕΣ προβλέπει 1,4 δις ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 12 και κάτι για την Νότια Κορέα δεν εντοπίστηκαν τομεί που θα επηρεαστούν αρνητικά από τις ΕΣΕ. Περίπτωση όμως που υπάρξει σοβαρή απειλή για κάποιου τομεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργοποιήσει πάρα αυτέ τι διαδικασίε ρήτρε διασφάλιση που προβλέπονται στη συμφωνία. Αν περαστεί ανάγκη, υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογή των ε, μέτρων στήριξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, η ΣΕΣ περιλαμβάνει φιλόδοξου δεσμού που υπερβαίνουν ακόμη και του κανόνε τη ΠΟΕ. Επίση, κανένα στοιχείο τη ΣΕΣ δεν έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, θέλουμε διάλογο και συνεργασία και ανταλλαγή ε, πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Θέλουμε να προωθήσουμε ενεργά την ε, σύμβαση της UNESCO του 2005 για την πράσπιση της πολιτιστικής ε, ποικιλομορφία και του πολιτιστικού πλούτου. Μετά από διαπραγματεύσεις με την Νότια Κορέα, καταλήξαμε σε διάφορες τροπολογίες της ΣΕΣ και των κανόνων της. Οι αλλαγές αυτές επιφέρουν μία πλούστευση μετά από ρητή αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα κάποιοι αυστηροί κανόνε διατηρήθηκαν για του ευαίσθητου τομεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία νέων ε, ευκαιριών ε, πρόσβαση στην αγορά των ευρωπαϊκών απορροκυρευτικών προϊόντων στη Νότια Κορέα. Και με εξαίρεση τα τρία πιο σημαντικά προϊόντα, την ντομάτα, το ε, τα πορτοκάλια και το κορεατικό κίτρο, ε, εσπεριδοειδή, ε, είχαμε άριστα δασμών και σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα για κάποιο τομέα υπάρχει ρήτρα διασφάλισης. Αυτή η ρήτρα διασφάλισης μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη θέση ισχύ της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Θα παρακολουθήσουμε τις τον αντίκτυπο των επιπτώσεων στις αγορές για να δούμε αν χρειάζεται η εφαρμογή της ρήτρα διασφάλισης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική ρήτρα επιστροφής δασμών. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη, τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών από την Νότια Κορέα. Η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία εξέφρασε κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά την ρήτρα για την ε, επιστροφή δασμών της ΣΕΣ. Αυτή τη στιγμή όμως ούτως ή άλλως ε, τη ρήτρα αυτή την χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς και οι Νοτιοκορεάτες. Η ΣΕΣ δεν προβλέπει νέα προνόμια και οι, επιπτώσεις, ε, οι οικονομικές επιπτώσεις των, της επιστροφής δασμών είναι μικρή. Ένα όγδο των, του συνολικού ποσού. Και μάλιστα από τη στιγμή που το εμπόριο θα αυξηθεί, η ρήτρα της επιστροφής της δεν θα έχει σημαντική επιρροή. Βέβαια, η εφαρμογή της ΣΕΣ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας και γι' αυτό η ΣΕΣ περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό άμεσης επίλυσης των διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσετε στενά την ε, υλοποίηση των υποχρεώσεων τη Νότια Κορέα και δεν θα διστάσει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό απειλήση διαφορών αν χρειαστεί. Η ΣΕΣ προάγει και τον σεβασμό του περιβάλλοντο και των εργασιακών δικαιωμάτων και περιλαμβάνει δεσμεύσει για την εφαρμογή πολλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Στόχο των δεσμεύσεων αυτών ε, είναι να εξασφαλιστεί προστασία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Επίση, έχουμε και ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση τη εφαρμογή συμφωνία αυτή με συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, επιχειρησιακών κύκλων, συνδικάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα εξέτασαν και την πιθανότητα προσαρμογή του συστήματο ε, κατάργηση των δασμών, κάτι που προποθέτει μεταξύ άλλων ότι τα προϊόντα που ταξινομούνται στα 3 και 5 χρόνια θα υποβάλλονται σε 4 και 6 περικοπέ δασμών, ώστε οι δασμοί να καταργηθούν ένα χρόνο αργότερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Βέβαια, αυτό μπορεί να μας δημιουργεί κάποια μικρά, μικρές απώλειες, αλλά νομίζω ότι έτσι λαμβάνονται υπόψη η ευαισθησία συγκεκριμένων τομέων. Άλλωστε, η Νότια Κορέα έδειξε την ετοιμότητα συμφωνία με τι αλλαγέ αυτέ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ευαίσθητοι τομεί και των δύο πλευρών. Σα ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θα περάσουμε στους αγορητές εκ μέρους των ομάδων, καταρχήν για δύο λεπτά και εκ μέρους του ΕΛΚ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στα νέα, νέα σας καθήκοντα. Ε, λαμβάνετε, αναλάβατε καθήκοντα σε ταραγμένα τραγμένες εποχές. Σας εύχομαι καλή τύχη. Για τη συμφωνία αυτή υπάρχουν ε, πολλά ωφέλη για την Ευρώπη. Είναι όμως μια ατυχή συμφωνία για την αυτοκινητομηχανία, όπως είπε ο Ντάνιελ Κάσπαρη. Κοιτάξτε τα νούμερα. Επίτροπε, για κάθε αυτοκίνητο που εξάγουμε εμεί από την Ευρώπη προς την Νότια Κορέα, 15 ξανάρχονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, 1 προς 15 είναι ο λόγος λοιπόν. Και αυτό βέβαια λόγω των μη δασμολογικών φραγμών ε, που ε, υπάρχουν για τις ε, εισαγωγές προς την Νότια Κορέα. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχει πια παραγωγή στην Ευρώπη, στην Αμβέρσα συγκεκριμένα, και να μεταφερθεί στην Νότια Κορέα η παραγωγή. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, ε, Επίτροπε. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε αυτό το πρόβλημα γιατί ε, επωφελείται γενικότερα η οικονομία της Ευρώπης. Πρέπει να βοηθήσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας και να αναφερθώ στη ρήτρα διασφάλισης. Πραγματικά θέλουμε να γίνει μια εισβάθος έρευνα του αντικτύπου αυτής της ε, συμφωνίας για την αυτοκινητομηχανία, να δούμε ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία ε, που είναι πάρα πολύ ανισχυτικά και η κυβέρνηση των ΗΠΑ βεβαίως διαπραγματεύεται ε, με την Νότια Κορέα μια παρόμοια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Να μην ξεχνάμε κύριε Επίτροπε ότι η αυτοκινητομηχανία είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος οικονομικός κλάδος κλάδος της ε, Ευρώπης με εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Δεν μπορούμε να χάσουμε και άλλες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να σας ζητήσουμε περαιτέρω εγγυήσεις ε, που θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και για τρία λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι αυτή η ΣΕΣ με την Κορέα είναι σημαντική για τρεις λόγους. Πρώτον, όπως είπατε, ε, μόνο ωφέλη δίνει ε, και για την Κορέα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους καταναλωτές, για τις θέσεις εργασίας και έχει και τη δυνατότητα να προσθέσει 19 δις στο εμπόριο, στην εμπορική ροή με την Κορέα. Δεύτερον, με τη συζήτηση που κάνουμε και δεδομένη της παγκόσμιας ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι θετικό παράδειγμα. Αν δύο μεγάλες οικονομίες όπως αυτές οι δύο μπορούν να συμφωνήσουν σε μία ΣΕΣ, αυτό δίνει όθηση και με άλλου εταίρου. Η Ιαπωνία ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο τώρα να έχει τέτοιου είδου ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι πριν από λίγα χρόνια και αυτό εν μέρη έχει να κάνει και με τη συμφωνία με την Κορέα. Από την άλλη πλευρά βέβαια οι Κορεάτες ε, τώρα ε, θέλουν πάλι να ε, ε, προωθήσουν και σχέσεις με τις ε, αργότερα. Είναι σημαντικό και για την Ευρώπη γιατί πολλές από τις αιτήσει, τα αιτήματα που εκφράζονται στην έκθεση προωθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω δύο-τρία παραδείγματα. Στην έκθεσή μου αναφέρομαι ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη πρόσβαση στην γεωργική αγορά της Κορέας. Η ε, γεωργικοί δασμοί θα μειωθούν 75% για 7 χρόνια που θα ισχύσει η συμφωνία. Ε, θέλουμε γεωγραφικούς, ε, θέλουμε προστασία ορισμένων προϊόντων μας και θα προστατεύονται όπως το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης το whisky 137.000 Ήδη ε, είναι πολύ μεγάλες οι πωλήσει και θα αυξηθούν μέσα από αυτή τη ΣΕΣ. Ε, θέλουμε οι μη τα μη δασμολογικά εμπόδια να αντιμετωπιστούν και αυτό θα ωφελήσει και την αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα εμπορικά και περιβαλλοντικά προϊόντα με αυτή την ΣΕΣ σε αυτό το τομέα εμπορεύματα και υπηρεσίες ε, μετά από τρία χρόνια θα, ε, τα προϊόντα μα θα μπορούν χωρίς δασμούς να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Το ίδιο θα ισχύσει και αντίστροφα. Ω Κοινοβούλιο θέλουμε ε, βελτιωμένα κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα. πρότυπα. Οι Κορεάτες μετά την ε, ΣΕΣ είπαν ότι θα προσχωρήσουν σε συμβάσει του ILO και θα ε, ε, υπάρξει δυνατότητα μετά από τη συμφωνία οι εταίροι στην Κορέα να ε, επιφέρουν και στον εργατικό τομέα, στην εργασία βελτιώσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι τέλεια συμφωνία. Όχι, προφανώς υπάρχουν πράγματα που δεν τα θέλουμε μέσα εκεί. Όμως στις, στις διαπραγματεύσεις έχουμε δούνε και λαβήν. Είναι σημαντική όμω η συμφωνία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κορέα και για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, και να την υπογράψουμε. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των φιλελευθέρων, για τρία λεπτά, το λόγο. κύριο Σερινάλντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, αυτό είναι ένα κλασικό θέμα στο οποίο παίζεται η φήμη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ε, Ευρωπαίους βιομηχανούς και καταναλωτές. Μία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών φαίνεται ότι είναι μια καλή είδηση. Πολύ περισσότερο όταν αντιπροσωπεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση την πρώτη επιτυχία της διμερούς εμπορικής πολιτικής μετά από μερικά χρόνια απογοητεύσεων. Ίσως γι' αυτό υπήρξε μια κάποια βιασύνη στην ε, ε, ε, μονογράφηση της συμφωνίας και ίσως υπήρξε ένας πειρασμός τέτοιος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλήξει η συμφωνία πάση θυσία. αν όμως η συμφωνία αυτή εφαρμοστεί αποτελεί μια αυτοκτονία για τη βιομηχανία. και αυτό αυτό θα αποτελέσει μια, ένα προηγούμενο και για τους άλλους εμπορικούς μας εταίρους. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε σκληρά, όμως όπως λένε στην Κορέα ε, ακόμα και οι πιο ε, καλοί κάνουν λάθη. Ε, η Κομισιόν έχει το καθήκον να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των παραγωγών, των καταναλωτών, ε, των εργαζόμενων και ε, πολλές φορές ε, ε, αυτά μέσα σε μια διαπραγμάτευση που κατακρίθηκε για έλλειψη διαφάνειας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από όλους μας μια πολιτική ευαισθησία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πάει άσχημα και είναι ε, περί ε, είναι άχρηστο ε, να επιδοτούν ε, σε κάποια κράτη-μέλη οι την αυτοκινοβιχαρία και από την άλλη μεριά να δίνουμε επιδοτήσεις με τον τρόπο αυτό στην αυτοκινοβιχανία της Νότιας Κορέας. Όλες αυτές οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν, η προστασία γεωγραφικών ονομασιών κλπ. Ε, όλα αυτά είναι θετικά. Αλλά μην ξεχνάμε τι γίνεται και στι ΗΠΑ, όπου η συμφωνία με την Κορέα εκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια και κάποιοι θέλουν να ανοίξουν και το κεφάλαιο τη αυτοκινητοφωνία. Η ερώτηση προ την Κομισιόν είναι η εξή. Το κείμενο τη συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει ένα πακέτο ε, συνολικό που θα περιλαμβάνει τρει πράξει. Την συμφωνία αυτή, τα εφαρμοστικά μέτρα, ιδιαίτερα για το duty drawback και τον κανονισμό για την ρήτρα διασφάλιση. Και ε, ενδεχομένω προσθέτω και την ε, πρόσβαση στο Ταμείο ε, Προσαρμογής για τους τομείς που θα πληγούν από αυτή τη συμφωνία. Όλα αυτά τα χαρτιά πρέπει να τα δούμε μαζί ε, και πρέπει να δούμε το, στα πλαίσια του κλίματος της συναπόφασης που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας να μην ε, ε, ε, αγνοηθεί το θέμα της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για την οποία θα πρέπει να, να εργαστούμε από κοινού. Για τρία λεπτά εκ μέρους των Πρασίνων το λόγο κύριο Ζαντό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι υπάρχει κάποια καινοτομία με τη νέα συμφωνία. Καινοτομία με τη νέα συμφωνία, αλλά τα λόγια είναι παρόμοια με αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμή. Και πρώτη φορά βλέπουμε στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων υπάρχουν, ότι υπάρχουν και κάποιοι χαμένοι. Το παραδεχόμαστε, αλλά στα πλαίσια μια εμπορική συμφωνία με τρίτους. Δεν είναι στα πλαίσια τη στρατηγική τη Λισαβόνα, δεν είναι στα πλαίσια τη βιομηχανική πολιτική που επιλέξαμε ποιοι θα είναι χαμένοι στην Ευρώπη ενό εμπορικού ανοίγματο προ την Νότια Κορέα. Καινοτομή λοιπόν η συμφωνία αυτή, γιατί συνήθω μία εμπορική συμφωνία ε, χαροποιεί τη βιομηχανία και δυσαρεστεί τη γεωργία. Εδώ το αντίθετο συμβαίνει. Σημαντική κλάδοι της βιομηχανίας παραπονιούνται για τις επιλογές της Ευρώπης. Καινοτομή λοιπόν η νέα συμφωνία γιατί μας αναφέρατε 1,6 δις μείωση των τελωνιακών δασμών στην νοτιοκορεατική αγορά. Τι σημαίνει αυτό το αριθμητικό στοιχείο. Εγώ εκλέγομαι στην, σε μια δυτική περιφέρεια της Γαλλίας, στη Βρετάνη. Αν πάτε στη Βρετάνη, κύριε Ντεγκούχτ, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα με τα φύκια με την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα εξαιτίας της ε, χειροτροφίας. Και είπατε ότι χάρη στην Συμφωνία Ελεύθερου θα κερδίσουμε στη χειροτροφία μας, θα έχουμε κέρδη με την εξαγωγή χείρων. Αυτή η δυτικοποίηση όμως της χειροτροφίας θα οδηγήσει σε μείωση θέσεων απασχόλησης, σε μείωση προστιθέμενης αξίας, σε απώλεια τουρισμού. Άρα η Βρετάνη θα βγει χαμένη από τι ΣΕΣ. Μπορεί ε, με συνολικά ποσά σε γενικούς όρους να κερδίζουμε, αλλά συγκεκριμένες περιοχές χάνουν. Άλλη καινοτομία της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου είναι ότι για πρώτη φορά ζητούμε περιβαλλοντική εξαίρεση, παρέκκληση. Γιατί μας ε, πείστε το μυαλό λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο αναφυσβήτητος ε, ηγέτης και πρωτοστατής στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και εδώ έχουμε στις διαπραγματεύσεις με την Κορέα μια παρέκκληση από, τους, ε, από τις διατάξεις για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων γιατί το λόμπι της Ευρώπης ε, ήταν πολύ ισχυρό και τώρα χρειάζεται κάποιες παρεκκλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν έγιναν δεκτές θέσεις εντός. Για ακόμη μια φορά λοιπόν περισσότερα θα υποστούμε παρά θα κερδίσουμε στη βιομηχανική πολιτική μας ή στην στρατηγική για τις επιχειρήσεις και στις οικονομικές μας επιλογές. Μας υπενθυμίσατε τη στρατηγική της Λισαβόνας, την πράσινη οικονομία και την καινοτομία και δεν βλέπω που η νέα συμφωνία θα ευνοήσει αυτούς τους τομείς. Μπορεί στη θεωρία να μας τα λέτε όλα ωραία, αλλά όταν μιλούμε για, τις, ε, για τη φορολογία τη φορολογία άθρακα ή τη φορολογία Τόμπιν, Σα στοιχηματίζω, κύριε Δικούχτ, ότι πριν την εκπνοή τη θητεία σα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να λάβει θέση για το φόρο Τόμπιν, που είναι απαραίτητο εργαλείο για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σα ευχαριστώ, κύριε Ζαντό. Εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών τη Ευρώπη, για δύο λεπτά, το λόγο έχει ο κύριο Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, με αυτή την ευκαιρία να σα καλωσορίσω στο νέο νέα σα θέση και σας εύχομαι πολύ επιτυχή θητεία. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι είναι καλό που γίνεται απόψε αυτή η συζήτηση και βγαίνουν σοφώς κάποια πράγματα. Είναι αλήθεια ότι πήραν, τράβηξαν σε μάκρος οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι θα μπορέσει η Κομισιόν να ολοκληρώσει και να κλείσει το θέμα σύντομα. Είναι μεγάλο το όφελος και για την Ευρώπη και για την Κορέα από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες, τις ακούω, τις ακούσαμε και σήμερα, αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά νομίζω ότι αν εξαρτηθούμε από την αυτοκινητοβιομηχανία και επικεντρωθούμε στην υποστήριξή της μόνο, νομίζω ότι θα κάνουμε λάθος και δεν νομίζω ότι η General Motors θα είναι η πιο σημαντική στην περιοχή μου ισότιμη αφορά. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες, συμμερίζομαι τις ε, πραγματικές ανησυχίες πολλών, τις κατανοώ, αλλά νομίζω ότι οι ευκαιρίες ε, ε, ξεπερνούν κατά πολύ τις ανησυχίες. Δεν νομίζω ότι αν είμαστε συγκρατημένοι θα επιτύχουμε. Πρέπει να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, όχι τα αρνητικά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η συμφωνία αυτή έχει και πολιτικό περιεχόμενο, γιατί Προς της Νότιας Κορέας υπάρχει ένας επιθετικός εχθρός και αποστέλουμε μήνυμα και προς τα εκεί, ποιον στηρίζουμε δηλαδή. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, να καταρρύψουμε τα εμπόδια σε αυτή την περιοχή. Η συμφωνία θα δείξει ότι ε, υποβοηθούμε την πρόοδο. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην περιοχή εκείνη και γνωρίζω ότι οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή τάσσονται υπέρ της πρόοδου ε, Υπάρχει υποστήριξη ε, αν, ε, βορανότου αν πάτε σε μια περιοχή όπως την Κεσόν. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσουμε και εμείς. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πρώτον. Πώς η Κομισιόν βλέπει τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών και πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Πόσο γρήγορα δηλαδή θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον μηχανισμό αυτό σε περίπτωση σοβαρών στρεβλώσεων της αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Φερέιρα. Κύριε Επίτροπε, Πολλέ φορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάσαμε τι ολέθριε συνέπειε τη απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου για πολλού ε, οικονομικού τομεί και ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη-μέλη και για ε, περιοχέ που εξαρτώνται από του τομεί αυτού. Μιλήσαμε για την καταστροφή τη παραγωγική ε, δραστηριότητα και απόλυθες θέσεων ε, έχουμε πρόβλημα στη δημιουργία και κατανομή του πλούτου. Αυξάνεται η εξωτερική μας εξάρτηση και χρονίζουν οι ανισορροπίες των εμπορικών μας οζυγίων, ε, οδηγώντας μας σε μια οικονομική κοινωνική ύφεση. Παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα, έχουμε κοινωνικό ντάμπικ, οδηγούμε στην πτώχευση ε, εκατομμύρια μικροπαραγωγούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι συνέπειες της ε, προοδευτική απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου που οι υπέρμαχοί του δεν μπορούν να τις αγνοούν. Για παράδειγμα, η κλωστιφαντουργία και ο τομέα ένδυση πλήττονται από την συμφωνία αυτή και η Eurofund δίνει σενάρια μείωσης ε, των θέσεων ε, εργασιες 20 25% μέχρι το 2020 και μακροπρόθεσμα μέχρι και απώλεια 50% των θέσεων απασχόληση. Ακόμη και ο ηλεκτρονικός τομής και η παραγωγή ανταλλακτικών θα ε, πληγούν από τη συμφωνία αυτή. Τέτοιες καταγγελίες έχουμε ακούσει και απάντηση δεν λαμβάνουμε. Τι μέτρα θα ληφθούν για τη διαφύλαξη των ε, τομέων αυτών. Χρειαζόμαστε μέτρα που δεν θα πρέπει απλώς να μετριάζουν την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Τι μηχανισμούς διασφάλισης θα έχουμε ή αναχέτησης των ε, επιθετικών εξαγωγών, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μετακατάσταση επιχειρήσεων. Με πρότασή μας, ο προϋπολογισμός του 2010 προβλέπει νέα κατηγορία για τις δράσεις στην κλωστή φαντουργία και στον τομέα ένδυσης και υπόδεσης. Ποια είναι τα κλειδιά του νέου προγράμματος. Χρειαζόμαστε δίκαιες και ισότιμες οικονομικές σχέσεις που θα εξυπηρετούν τους φτωχούς πολίτες και χώρες και όχι κάποια λόμπι και ο, μήλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε η φόρα ανάπτυξη. Αυτή είναι η απέτηση των επερχόμενων γενεών και μια οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, ενεργειακή ορθολογικότητα που το φιλεύθερο μοντέλο όχι μόνο δεν εξασφαλίζει αλλά αντίθετα υποσκάπτει. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε το γύρο των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων με την κυρία Ρόσπαχ που θα μιλήσει για δύο λεπτά εκ μέρους της ελευθερίας, της, ε, της δημοκρατίας, ελευθερίας και δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Νότια Κορέα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και πραγματικά είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε εμπορικές συμφωνίες με την ε, Νότια Ασία. Πρέπει να συνδέσουμε όσο πιο πολύ τις χώρες αυτές με την Ευρώπη. Ε, φυσικά υπάρχει, υπήρχε για πολύ καιρό μια ανισορροπία στις εμπορικές συναλλαγές ε, με την Νότια Κορέα λόγω του προστατευτισμού της Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα πριν από μερικές δεκαετίες ε, άρχισε να αναπτύσσεται και εξελίχθηκε σε μια βιομηχανική κοινωνία. 80% του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Η χώρα είναι σήμερα η ενδέκατη μεγαλύτερη οικονομία ε, στον κόσμο και ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμμαχό μα σε διάφορους στρατηγικούς τομεί. Η πρόγνωση είναι ότι θα αποκτήσει όλο και πιο δεσπόζουσα θέση η χώρα αυτή στις, ε, στο, στο, στον τομέα της, των προϊόντων υψηλή τεχνολογία την επόμενη δεκαετία. Η Νότια Κορέα πρέπει να ανταγωνιστεί ε, με την Βόρεια Κορέα και την ε, Κίνα, που βεβαίως είναι ο μεγαλύτερος της ε, εμπορικός εταίρος. Η Κίνα έχει ανεξάρτητους πόρους και φθηνό εργατικό δυναμικό και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός ανταγωνιστής η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέτει απαιτήσει ποιοτικού χαρακτήρα ε, προς την ε, Νότια Κορέα. Και αυτό θα είναι κάτι το θετικό. αυτή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών όπως ακούσαμε, θα μειώσει τους δασμούς κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό φυσικά είναι πολύ ε, θετικό. Για μένα όμως ε, το ερώτημα είναι το κατά πόσον έχουν απελευθερωθεί αρκετά οι επιχειρήσεις της ε, Νότιας Κορέας και αν ε, μπορεί να τηρηθούν οι όροι της ε, συμφωνίας αυτής, διότι η Νότια Κορέα δίνει ακόμα επιδοτήσεις σε μεγάλους οικονομικούς κλάδους όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά. Το λόγο ο κύριος Πέτερ Σιάστηνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες είχαμε ε, αλλαγές και μεταβάσεις, ε, είχαμε τους επιτρόπους ε, για το διεθνές εμπόριο, είχαμε επίσης τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη Νέα Επιτροπή. Πάντα ετώνιζα σε ανώτατο επίπεδο ε, την ανάγκη βελτίωσης ε, της ΣΕΣ ε, με την Νότιο Κορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένα συμφέροντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυτοκίνητο βιομηχανία. για τη ρήτρα ασφάλισης, μη δασμολογικούς φραγμούς, αυτά ήταν θέματα τα οποία ετώνησα. Θα πρέπει να με περισσότερο την συμφωνία. Ακόμα και η ΕΠΑ ε, επιθυμεί τέτοια συμφωνία, ε, αλλά υπάρχουν παρόμοιες συνστάσεις από, από την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτή είναι πολύ σημαντική, είναι η πρώτη ΣΕΣΕ, είναι ένα υπόδειγμα, πρέπει να γίνει σωστά ε, και θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες του παιχνιδιού και για τους δύο. Μην με παρεξηγήσετε κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι σαφώς υπέρ της ΣΕΣΕ, κατανοώ το θετικό αντίκτυπό της στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ε, ότι όταν είναι μονόπλευρο το συγκριτικό πλεονέκτημα θα μειωθούν τα ωφέλη και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είναι αρνητική η εξέλιξη. Ε, η βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπιστεί καλύτερα στην Ευρώπη. Θα πρέπει ίσως ε, με το διατλαντικό εταίρο μας να ζητήσουμε κάποιες προσαρμογές που θα καλύψουν τις τεράστιες αυτές βιομηχανίες μας ε, για να βελτιωθεί η ΣΕΣ. Ε, συνολικά η ΣΕΣ θα πρέπει να είναι ε, επωφελής και για τις δύο πλευρές. Είναι δική μου ευθύνη και καθήκον να παρακολουθώ και να διασφαλίζω ότι οι εκλογείς, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν μια δίκαιη συμφωνία. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά το λόγο κύριο Σαρίφ. Μου τα γυαλιά, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Ήδη το Σεπτέμβριο συζητήσαμε στην Ολομέλεια την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Νοτιού Κορέα και μάλιστα πολλοί εκφράσαμε επιφυλάξει και φόβου για τι αρνητικέ συνέπειε τη συμφωνία αυτή, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε ότι τα στοιχεία θα μα δικαιώδαιναν. Το 21 Ιανουαρίου η Όπελ ανήγγειλε το κλείσιμο του εργαστασίου τη Αμβέρσα με μετακατάσταση στη Νότια Κορέα. Πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή είναι άσχετη με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Μάλλον όχι. Σίγουρα υπάρχει κάποια σχέση. Στην περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου οι, εργαζόμενοι πληρώνουν τα σπασμένα των λαθών των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξετάζει δεόντως τις συμφωνίες, των, των, συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών. Οι, άνθρωποι χάνουν τις, τη δουλειά τους και εμείς ε, θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι στο διεθνές εμπόριο υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι και χαμένοι θα είναι αυτοί γιατί αυτούς τους θυσιάζουμε στο βωμό του παγκόσμιου εμπορίου. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από σας κύριε Επίτροπε. Η Γενική Διεύθυνσή σας αξιολόγησε το, την επίπτωση συμφωνίας αυτή στην απασχόληση Ευρώπης. Γιατί ε, τα στοιχεία που μας δώσατε ότι θα έχουν 19 ε, εκατομμύρια ευρώ κέρδη η Ευρωπαίοι βιομήχανοι δεν ξέρω πού στηρίζεστε, γιατί δεν νομίζω ότι λήφθησαν υπόψη αρνητικέ ε, επιδράσει αυτή τη συμφωνία. Αναφέρθηκαν οι ρήτρε διασφάλιση και η επιστροφή ε, δασμών. Πρώτη φορά δίνουμε τέτοια προνόμια, ακόμη και σε αναπτυσσόμενε χώρε δεν ε, καταφεύγουμε στο μέτρο αυτό. Βέβαια είπατε ότι υπάρχει δυνατότητα εφαρμογή ρήτρε διασφάλιση. Για πρώτη φορά όμω, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτό το κείμενο με βάση τη συναπόφαση. Δεν νομίζω ότι ε, χρειάζονται βαλωματικά μέτρα για να διορθώσουμε το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια γνήσια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και μια πραγματική στρατηγική για το μέλλον των βιομηχανιών μας. Γιατί σε μια παγκόσμια κρίση και οξυμένη ε, σε ξημένο ανταγωνισμό θα πρέπει να έχουμε συντονισμένη εμπορική πολιτική ότι οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών να μην καταστρέφουν τι θέσει εργασία στην Ευρώπη. Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο περιμένουμε εξηγήσει είναι το θέμα του πρωτοκόλου για την πολιτιστική συνεργασία που περιλαμβάνει η συμφωνία. Πολλέ χώρε αντέδρασαν έντονα στι διαπραγματεύσει με την Νότια Κορέα που δεν έχει καν. Ε, προσυπογράψει την σύμβαση της UNESCO για την πρόθεση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Καταγγέλλω λοιπόν ακόμη και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πολιτιστικά θέματα. Τα πολιτιστικά θέματα είναι άσχετα με τα εμπορικά και θα πρέπει να τα διαπραγματευτεί ο αρμόδιος επίτροπος πολιτισμού, ώστε να μην γίνει ο πολιτισμός ένα στοιχείο ε, διαπραγμάτευση, να ήταν ένα κοινό εμπορικό αγαθό. Θα πρέπει επίση να ενημερώνεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι τρέχουσε διαπραγματεύσει σε όλα τα στάδια και για το περιεχόμενο τη διαπραγματευτική εντολή. Πέραν των δισταμένων απόψεων, χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόωρο στάδιο, ώστε να έχουμε εμπεριστατωμένη γνώμη για τη στρατηγική σα. Περιμένουμε συνεργασία μαζί σα και με του αρμόδιου άλλου επιτρόπου γιατί όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε μια πιο γνήσια κοινοτική εμπορική πολιτική που θα είναι όμως και πιο δίκαιη. Ευχαριστώ Καντέρ. Μιλάς πολύ γρήγορα και δεν σε προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Μου κάνουν συνέχεια νοήματα ότι δεν μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Τρέχεις από λιβόλο Και έχεις και πολύ περισσότερα λεπτά και σε αφήνω και παραπάνω. Αλλά είσαι με δραλιοβόλο. Δεν σε προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Μόνο οι Γάλλοι σε καταλαβαίνουν έτσι πως μιλάς. Το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόσα, η Μπαλσέλης, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε Ντεχούκτε, Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση ελευθέρωσης συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Κορέα είναι σημαντική συμφωνία και αφορά ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή αυτοκτοβιομηχανία και την κλώστο υφαντουργία που οι δύο αυτοί κλάδοι εξέφρασαν ανησυχίε για συγκεκριμένα θέματα όπως το σύστημα drawback και τη ρήτρα διασφάλισης. Επίσης, ε, η TUC, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, ε, επέκρινε αυτή τη ε, συμφωνία. Η Νότια Κορέα δεν έχει επικυρώσει καμία από τις θεμελιώδεις συνθήκες και συμβάσεις του ILO. Η Νότια Κορέα συνεχώς καταβιάζει και παραβιάζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Επιπλέον, ξέρουμε ότι για αυτή την συμφωνία υπήρχε σαφής διάσταση απόψεων μεταξύ των επιτρόπων και επίσης ανάμεσα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Ταξούτ και στη Γενική Διεύθυνση Τρέιτ σχετικά με το σύστημα ε, επιστροφής δασμών. Ε, ε κατά την ταξούντ αυτό δημιουργεί ε, οικονομικές στρεβλώσεις γιατί είναι μια έμεση επιδότηση και αυτό δημιουργεί σαφές ε, ε, πλεονέκτημα κατά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπέρ της ε, κορεατικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο ίδιος ο οργανισμός πρόθεσης των επενδύσεων ε, της Νότιας Κορέας ε, υπολόγισε ότι το πλεονέκτημα αυτό είναι περίπου 1.300 ευρώ ένα αυτοκίνητο. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι δίκαια συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια επικαιροποιημένη ε, μελέτη ε, αντικτύπου ε, της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει Ζαλεύσκη. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα εξετάζουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία που, κανονικά θα γίνει υπόδειγμα και συμφωνιών με άλλες ε, χώρες της από ή της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας. Γι' αυτό χρειάζεται διεξοδική ανάλυση και δεν θα πρέπει να δράσουμε υποπίεση χρόνου. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη και στην πολιτική σταθεροποίηση, αλλά θέλουμε έναν ανταγωνισμό που θα είναι ισορροπημένος και θα στηρίζεται στην τεχνολογία ή στο κόστος παραγωγής προϊόντων και δεν θα στηρίζει το ανταγωνισμός αυτός στην, στους δασμούς για τα πουλερικά, για παράδειγμα, ή για, για, για ορισμένα προϊόντα. Έχουμε ε, μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, οπότε θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για την κατάσταση στην Ευρώπη και επίσης να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όχι μόνο της αυτοκίνητο αλλά και της βιομηχανίας ηλεκτρικών ειδών και της κλωστοϊφαντουργίας. Υπάρχουν πολλοί τομεί που παραπονιούνται για τη συμφωνία αυτή, ακόμη και στην Πολωνία. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δράσουμε με τον εξή τρόπο. Καταρχήν, θα πρέπει να ενημερωθούμε διεξοδικά για τις συνέπειες της ε, συμφωνίας αυτής και να συνεργαστούμε με τους τομείς, όχι με αυτούς που είναι ικανοποιημένοι και θα βγουν κερδισμένοι από τη συμφωνία, αλλά και με τομείς που έχουν επιφυλάξεις για τη σύναψη της συμφωνίας. Και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μερόληπτη και αντικειμενική ανάλυση των επιπτώσεων της συμφωνίας αυτής. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ διεξοδικά και τις ρήτρες διασφάλισης. Να δούμε τι περιεχόμενο θα πρέπει να έχουν για να αποβεί ε, αμοιβαία επωφελής η συμφωνία αυτή και να μην ε, ωφελήσει μονομερό στην Νότια Κορέα. Επίσης δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε προσωρινά τη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε τη γνώση τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να πιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η συμφωνία αυτή είναι υποφελή για όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δημιουργεί ε, προνόμια και μεταχείριση διακριτική υπέρ τη Νοτιού Κορέα. Σα ευχαριστώ για δύο λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριο Βιτάλ Μορέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω στον αρμόδιο επίτροπο εμπορίου δύο ερωτήσεις για το νόημα αυτής της συμφωνίας για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την αναγγελία της στρατηγικής ε, για την ε, Παγκόσμια Ευρώπη του 2006 με στόχο την ε, ενίσχυση του, του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομικής στρατηγικής της Ένωσης αυτή είναι η πρώτη αλλά και μοναδική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που έχει διαπραγματευτεί αλλά ακόμη δεν έχει ε, επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικό εμπορικό εταίρο ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια πολύ διεξοδική αξιολόγηση για το κατά πόσο οι στόχοι του Global Europe έχουν υλοποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, ελάχιστα έχουν επιτευχθεί. Η ίδια η αξιοπιστία της εμπορικής ε, πολιτικής της Ένωσης διακυβεύεται στην συμφωνία με την Νότια Κορέα. Από την επικύρωση της ε, συμφωνίας αυτής θα εξαρτηθεί η ίδια η αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία αυτή είναι η διμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτης Χώρας. Η σύναψη πολυμερών συμφωνιών εμπορικών δυστυχώς ε, έχει περάσει δεύτερη μοίρα μπροστά στις διμερείς συμφωνίες. Ακόμη και οι περιφερειακές συμφωνίες έχουν επισκιαστεί από τις διμερείς. Με όλα αυτά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η διμερή συμφωνία ε, μαρτυρεί την προτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες και όχι για πολυμερείς. Και είμαστε καταδικασμένοι σε ισόβια ε, σύναψη διμερών συμφωνιών. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά το λόγο ο κύριος Ζάλμπα. Κύριε Επιτροπέ, η θέση του ΕΛΚ είναι απερίφαστη και σαφής ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε έθερμοι υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαπραγματεύεται εμπορικέ συμφωνίε και με άλλε χώρε, γιατί με αυτέ δημιουργούνται νέε ευκαιρίε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και νέε θέσει απασχόληση που τι χρειαζόμαστε σε, αυτό το, σε αυτή τη σοβαρότητα οικονομική κρίση που διανύουμε. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια σα, κύριε Επίτροπε, γιατί και κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό οι συμφωνίε αυτέ να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την, ε, και την αποφυγή άδικων ε, ρητρών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη συμφωνία μιας νέας γενιάς εμπορικών συμφωνιών που είναι πιο φιλόδοξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η σημασία τη συμφωνία αυτή. Είναι άσχετο αν η χώρα με την οποία συνάπτουμε τη συμφωνία είναι μικρή ή μεγάλη. Το θέμα είναι να μην αποδυναμώσουμε τη διαπραγματευτική μα ε, ισχύ σε μελλοντικέ μα εμπορικέ συμφωνίε με μεγαλύτερε χώρες και εμπορικού εταίρους. Δεν είμαστε κατά της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Νότια Κορέα. Θέλουμε όμως να εξεταστούν πιο διεξοδικά και αυστηρά κάποιοι παράγραφοι της συμφωνίας που κατά τη γνώμη μου δημιουργούν συγκριτικά μειονεκτήματα και αθέμητο ανταγωνισμό για ορισμένους βιομηχανικούς τομείς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευνοούν δυσανάλογα τους νοτιοκορεάτες παραγωγούς και κατασκευαστές. Γιατί λοιπόν η ρήτρα διασφάλισης για την επιστροφή των δασμών θα τεθεί σε ισχύ μετά από πέντε χρόνια. Μου είπατε ότι ο λόγος είναι ότι οι δασμοί για τα οχήματα θα εξαλειφθούν, θα καταργηθούν μετά από πέντε χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει ότι σε πέντε χρόνια θα καταργηθούν οι δασμοί για τα οχήματα με βάρος άνω των 5 τόνων. Παρ' όλα αυτά, για τα ελαφρότερα οχήματα κάτω των 5 τόνων, που είναι όλα σχεδόν τα συμβατικά οχήματα, ο δασμό του 10% θα εξαλειφθεί σε τρία χρόνια. Οπότε τι γίνεται με τη διετία που περισσεύει. Θέλουμε πιο διεξοδικές απαντήσεις για τις καινοτομίες της Νέας Συμφωνίας. Τι νόημα έχει να διορθώνουμε τα προβλήματα κατόπιν εορτής, ενώ η ρήτρα διασφάλισης ε, προσπαθεί να προλάβει τις αρνητικές συνέπειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάλμπα. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ΣΕΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνάπτονται με χώρες που σέβονται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι κανόνες του Διεθνούς Γραφείου Εμπορίου. Είναι πολύ καλές οι αναφορές στα εργασιακά θέματα, αλλά δεν είναι πλήρης. Πολλές φορές συνδικαλιστικά δικαιώματα παραδιάζονται, συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται σωστά, όπως και το δικαίωμα ε, του, των ε, συνεργασιών παραβιάζεται στη χώρα αυτή. Επίσης αναμένονται προβλήματα όπως αναφέρθηκε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, τα προβλήματα της Όπελ τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Επίσης, πολλές φορές τα προβλήματα δεν παρουσιάζονται ε, σωστά. Τα προβλήματα της μετεγκατάστασης ε, είναι πολύ σοβαρότερα. Ποιος ωφελείται. Δεν... Ε, ε, λύνονται τα προβλήματα αυτά από την ΣΕΣ. Επίσης, ο ναυπηγικός τομέας είναι πολύ σημαντικό στην Κορέα. Ο στόχος είναι το 90% ε, των ναυπηγουμένων σκαφών να προέρχονται ε, από την Κορέα, πράγμα πολύ ε, ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους απασχολουμένους στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά, για δύο λεπτά ο κύριος Λάνγε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Λάγκε. Ο συνάδελφος θέλει να κάνει μια ερώτηση στην κυρία Ρέγνερ. Δέχεστε να σας κάνει ο συνάδελφος μια ερώτηση η κυρία Ρέγνερ. Κυρία Ρέγνερ μετά από την εφαρμογή της διαδικασίας της ε, μπλε κάρτας, εγώ είμαι κατά της διαδικασίας ε, αυτής, ε, αλλά θα κάνω μια εξαίρεση. Ε, υπάρχει συνάδελφος που επιθυμεί να σας κάνει ερώτηση. Το δέχεστε? Το δέχετε. Κάντε παρακαλώ την ερώτησή σας στον 30 δευτερόλεπτο, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε για την ευκαιρία που μου δίνετε. Αναφερθήκατε στην ε, Opel και στην Αμβέρσα. Ε, συμφωνείτε ότι η εταιρεία Opel εδώ και μήνες έχει μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και η Opel θα μπορούσε να παραγάγει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι κάνει και ότι η κακή οικονομική κατάσταση της Opel ε, προκλήθηκε από, δεν προκλήθηκε από μια ΣΕΣ η οποία δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή. Επιθυμείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Ένα λεπτό. Αλήθεια είναι βεβαίως ε, υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εδώ, σίγουρα. Αλλά υπάρχει μια συμφωνία ΔΕΛΤΑ από τη διοίκηση της εταιρεία και από τη διοίκηση παραβιάστηκε, από την διοίκηση Ορίλη και είχε διασφαλιστεί στην Opel Αμβέρσα ότι εκεί θα παράγονται, θα κατασκευάζονται μοντέλα SUV που δεν παράγονται στην Αμβέρσα αλλά κατασκευάζονται στην Κορέα. Ως εκ τούτου Πρόκειται για μετεγκατάσταση ε, της Opel Amversa προς την Νότια Κορέα. και προχωρούμε στην κανονική διαδικασία Τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Λάνγκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, τρεις ερωτήσεις θα σας απευθύνω. Πρώτη ερώτηση. Χρειαζόμαστε δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού. Βλέπω ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων περιορίζονται στη Νότια Κορέα. Άρα είναι αθέμητες οι συνθήκες ανταγωνισμού εκεί. Για παράδειγμα, το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο ποινικό κώδικα στην παράγραφο 314 στην Νότια Κορέα προβλέπει ποινικό αδίκημα την ε, διατάραξη της τάξης της επιχειρήσης. Αυτό υπάρχει για να ε, εμποδίζονται οι απεργίες και ε, να περιορίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στην Ζουγζουγ, για παράδειγμα, και διαρωτώ με γιατί πρέπει να συνάπτονται ΣΕΣ με χώρες που έχουν ε, μεγάλα προβλήματα όπως η Νότια Κορέα και η Κολομβία με την, τον ILO. Με αυτή τη ΣΕΣ πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχουν συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού και περιορισμός των, ε, εργατικών, των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επίσης, αναφέρθηκαν από πολλούς τα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, σωστές ρήτρες ασφαλείας. Και αν το προσέξουμε, υπάρχουν κάποιε γενικέ ρήτρε ασφαλεία όταν πρόκειται για μεγάλη ε, διαστρέβλωση ε, του εμπορίου ή υπάρχει ρήτρα ασφαλεία για το σύστημα επιστροφή των δασμών. Δεν μπορώ να το καταλάβω. μπορείτε με απλά λόγια να μου εξηγήσετε αυτή την ρήτρα ασφαλεία και συγκεκριμένα πώ ενεργοποιείται, από ποιον και πότε. Τρίτη ερώτηση. Ε, με την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε νέα ε, βάση ε, συμβατική για τη συνεργασία μας. Οι ρήτρε ασφαλείας και η εφαρμογή τους θα αποφασίζονται με συναπόφαση. Μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο όταν θα μπορέσει να έχει ασκήσει τα δικαιώματά του το Κοινοβούλιο και όταν θα έχει εγκριθεί η, η, η ρήτρα ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είμαι σίγουρη, ότι οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών δεν συνάπτονται για ιδεολογικού λόγου, αλλά γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι αποτελέσματα θα έχουν στι ε, κοινωνίε μα. Μιλάω για τι κοινωνικέ και οικονομικέ επιπτώσει. Αναφερθήκατε σε κάποιε μελέτε αντικτύπου. Εγώ όμω ποτέ δεν ε, διάβασα καμία ε, μελέτη που να αναλύει ανακλάδο κλάδο οικονομικό, βιομηχανία, τι αποτελέσματα θα έχει μια τέτοια συμφωνία στην απασχόληση. Έγινε λόγο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο καθένας ε, κοιτάζει την περιοχή του, κοιτάζει τη χώρα του και ξέρουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσεις. Ε, θα κλείσει το εργοστάσιο ε, της Όπελ στην Αμβέρσα και τα συνδικάτα που λειτουργούν στην Αμβέρσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πεπισμένα ότι η συμφωνία αυτή είναι η υποκείμενη αιτία της μετεγκατάστασης της ΟΠΕΛ. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Έχετε δει καμία ε, σαφή μελέτη αντικτύπου ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η συμφωνία στην απασχόληση ανατομέα. Αν δεν υπάρχει τέτοια μελέτη θα ήθελα να σας ε, ε παροτρύνω να ε, παραγγείλετε μια τέτοια μελέτη. Χρειάζεται μια τέτοια μελέτη το Κοινοβούλιο για να ασκήσει τις εξουσίες του. Δεύτερον, έχετε σαν σκοπό να πραγματοποιήσετε στο μέλλον ε, τέτοιες μελέτες σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις τέτοιων συμφωνιών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο κύριος Ρινάλντι θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Δέχεστε την ε, ερώτηση αυτή. Έχετε το λόγο κύριε Ρινάλτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να επωφεληθώ από την διαδικασία Catch the Eye για να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση προς τον Επίτροπο. Τότε μη σηκώνετε την πλακάρτα, σας, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα όντως στη διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτος, ο κύριος είναι ο Σον Κέλλη. Ένα λεπτό ο καθένας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα υπάρξουν ε, κερδισμένοι και χαμένοι με την ε, σύμφωνία αυτή. Η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να είναι από τους χαμένους. Η ερώτηση είναι, θα αυξηθεί η ζήτηση για αυτοκίνητα τα επόμενα 30-40 χρόνια και ίσως εκεί υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες. Αλλά συνολικά μίλησε ο, ο Επίτροπος για ένα όφελος 19 δισεκατομμύρια για την ευρωπαϊκή οικονομία και 12 κάτι για την κορεατική. Ε, και ότι αυτό είναι μια καλή συμφωνία κατά συνέπεια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια ψυχολογική διάσταση ότι απλώνουμε το χέρι προς τους εταίρους μας αυτούς σε μια περιοχή όμως του κόσμου που υπονόμευσε την συμφωνία της στην Κοπεχάγη. Ε, τελείωσε το λεπτό σας, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ντέση. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή η συμφωνία με την Κορέα είναι η πρώτη που θα εφαρμόσει ε, την στρατηγική Global Europe και πρέπει να είναι υποδειγματική γιατί δημιουργεί προηγούμενο. Όμως διαπιστώνουμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα πρόβλημα ενημέρωσης ε, του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ρήτρα διασφάλισης, ένα πρόβλημα μεθόδου γιατί ε, τίθεται σε, προφο... σε προσωρινή ισχύ η συμφωνία χωρίς να περιμένουμε τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, ένα πρόβλημα διαφάνειας, όπως είπε και ο κύριος Ρινάλντι, γιατί μέσω της ρήτας drawback θα ε, είναι σαν να συνάπτουμε έμεσα συμφωνία με την Κίνα και υπάρχει και ένα θέμα ε, συνέπειας με τις ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας φιλοδοξίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι διαπραγματεύονται κοινωνικές ρήτρες στις συμφωνίες τους με την Κορέα. Και στην οικονομική στιγμή που βρισκόμαστε, με την αυτοκινητομηχανία... Κόβεται το μικρόφωνο. Το λόγο έχει ο κύριος Ρινάλντι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ε, συμπληρωματική ερώτηση, λοιπόν, προς τον Επίτροπο. Καταλάβαμε ότι δεν έχουμε σαφές πλαίσιο όσον αφορά τη διαδικασία ε, ενδεχομένης επικύρωσης από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ποια είναι όμως η πλειοψηφία που θα πρέπει στο Συμβούλιο να επιτευχθεί ε, για να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, χρειάζεται συνένεση. Δεν το έχω καταλάβει αυτό και είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η νομική βάση. Προσθέτω ότι βρίσκω περίεργο το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης. Γίνω... Υπάρχουν πολλές ε, ανησυχητικές ε, ε, πτυχές και καλό την ε, Κομισιόν να επεξεργαστεί όλα αυτά τα θέματα μαζί μας. Ε, υπάρχει μια άλλη κορεατική παροιμία που λέει «Ψάξε το δρόμο ακόμα και αν τον ξέρεις» και σας ευχαριστώ την προσοχή σε αυτό. Ε, το λόγο έχει ο κ. Σικέσκη τώρα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η ΣΕΣ με την Νότιο Κορέα φαίνεται πολύ καλή κίνηση. Μιλάμε για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα αυξήσει το εμπόριο μεταξύ των δύο μερών. Ως αποτέλεσμα της απάλληψης των κορεατικών δασμών ε, ύψους 1,6 δις και ως αποτέλεσμα της εξάλληψης ευρωπαϊκών δασμών θα υπάρξει αύξηση εμπορίου ε, αγαθών και υπηρεσιών. Ε, επίσης, η ΣΕΣ θα συμβάλλει στην αύξηση της ε, διαφάνειας. Στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερα πιστοποιητικά, καλύτερης ποιότητας. Είναι πολύ σημαντική η επιρροή αυτή τη συμφωνία στην οικονομία, γιατί θα επιτρέψει τη σύντομη άμεση οικονομική ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Δυστυχώ, εξαντλήθηκε ο χρόνο τη κυρία Σικέρσκη και διακόπτει ο πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε την διαδικασία Catch και θα ολοκληρώσουμε με την δευτερολογία του Επιτρόπου που θα σχολιάσει τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Κύριε Τεχούχτα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, γιατί πολλές ερωτήσεις ε, έχουν ε, αναφερθεί σε αυτήν. Προφανώς για πρώτη φορά αφενός το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συγκατατεθεί ε, για τη συμφωνία και δεύτερον οι ρήτρες ασφαλείας θα πρέπει να εγκριθούν με συναπόφαση και αυτό έχει νομίζω επιπτώσεις για τις σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Οι ρήτρε διασφάλισης ε, είναι οι προτάσεις της Κομισιόν που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες και θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πολύ σύντομα και προφανώς ε, εκεί θα ακολουθηθεί η διαδικασία συναπόφασης. Γιατί λοιπόν οι τόσες παρατηρήσεις, ερωτήσεις, αμφιβολίες σε σχέση με τις ρήτρες διασφάλισης. Θα είναι ρήτρες διασφάλισης που θα τύχουν τη σύμφωνη γνώμη σας, αφού μιλάμε για συναπόφαση. Δεν βλέπω γιατί υπάρχει λόγος για τόση ανησυχία από την πλευρά σας και την ε, επικύρωση. Η επικύρωση από το Κοινοβούλιο συνεπάγεται και προϋποθέτει συζήτηση στην Επιτροπή σας. Είπα και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι δεν πρόκειται να κάνω πρόταση για πρόορη εφαρμογή των διατάξεων εκτός και αν το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί επί της συνθήκης συνολικά είτε πρόκειται για την επίσημη επικύρωση από το Κοινοβούλιο ή αν θα προβλεφθεί άλλη διαδικασία ε, που θα θεσπίσουμε μεταξύ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ανοιχτό, μπορεί να συζητηθεί. Εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να αποφανθεί πολιτικά επί της, συνθήκης, επί της συμφωνίας πριν ε, υπάρξει πρόταση για ε, ε, νωρίτερη εφαρμογή. Ένα άλλο θέμα. Είναι μεικτή συμφωνία αυτή, είναι μια συμφωνία που αφορά μόνο τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Η νομική υπηρεσία τώρα ετοιμάζει την σχετική γνωμοδότηση, αλλά μπορεί στο τέλος να πρέπει να θεωρηθεί μεικτή συμφωνία που σημαίνει ότι και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να επικυρώσουν και απαντώντας τον Νικολό Ρινάλδη μπορεί να έχει αυτό ε, επιπτώσεις στη διαδικασία ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Αυτά για τη διαδικασία και θα έχετε όλες τις δυνατότητες να αποφανθείτε και εμείς ε, σχολαστικά θα, θα ε, ε, ακολουθήσουμε τις απόψεις σας, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα, η ερώτηση για την ε, Όπελ και την Αμβέρσα, ε, αυτό είναι ένα θέμα βελγικό, αλλά και άλλα κράτη-μέλη ανησυχούν. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Λέτε, ας πούμε, αν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ με την Νότια Κορέα και το γεγονός ότι έκλεισε εδώ ένα εργοστάσιο της Όπελ στην Ευρώπη. Η Όπελ το 2009 ε, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 20% το παραγωγικό δυναμικό της στην Ευρώπη. και βέβαια θα μπορούσε να γίνει βέβαια διατηρώντας όλα τα εργοστάσια ανοιχτά. Αυτή όμως ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τη διοίκηση της Όπελ. Παράλληλα όμως η απόφαση η εισαγωγή SUV από την Νότιο Κορέα προήλθε ε, έλαβε χώρα μετά την συμφωνία αλλά πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις ΣΕΣ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το χρονικό ορίζοντα, η... δεν είναι σωστή η ισχυρισμή της κυρίας ε, ε, Βαν Μπρέμπτ και άλλων. Είπατε ότι υπογράφει η συμφωνία με την Νότια Κορέα. Θα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε αυτό που λέτε και να πούμε ότι κάποια κράτη-μέλη συμφώνησαν με την ΣΕΣ με την προϋπόθεση ότι θα εγνώριζαν τι θα συνέβαινε με την Όπελ. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να πούμε ότι, ε, γιατί είπατε εσείς ότι η Νότιος Κορέα ε, εξάγει 15 φορές περισσότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη ε, από ό,τι αντίστροφα. Εδώ υπάρχει ένα μαθηματικό σφάλμα. 730.000 εξάγονται από την ε, Ευρώπη στην Κορέα και 440.000 από την Κορέα στην Ευρώπη. Ούτε το επιχείρημα είναι σωστό γιατί προϋποθέτει ότι οι αγορές είναι ίσου μεγέθους, ενώ αν συγκριθούν διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ μικρότερη η νοτιοκορεατική αγορά από την ευρωπαϊκή. Δηλαδή συγκρίνεται ανώμια μεγέθη. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τη δίσδυση στην αγορά, δεν έχουμε το ίδιο ποσοστό ε, Ευρώπη προς Κορέα και αντίστροφα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πολύ σημαντικότερο να εκτιμήσουμε την κατάσταση στις αγορές και να πούμε ότι οι νοτιοκορεάτες παραγωγή πρόσφατα άνοιξαν μεγάλα εργοστάσια. Στην Τσεχία, για παράδειγμα. Το δεύτερο δεν θυμάμαι που είναι, στην Ευρώπη πάντως και στη Σλοβακία. Που αυτό σημαίνει ότι και τα δύο έχουν δυναμικό παραγωγής 500.000 αυτοκίνητα ετησίως. Έτσι λοιπόν στο μέλλον θα, παράγονται, θα κατασκευάζονται νοτιοκορεατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη και θα είναι ως επιτοπλίστων τα ε, αυτοκίνητα αυτά που θα μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας βλέπουμε λοιπόν μια μετατόπιση προς τις μεγάλες αγορές όπου θα λαμβάνουν χώρα και οι πωλήσει, ε, οι μεγαλύτερες πωλήσει των αυτοκινήτων. Ε, βέβαια είναι πολύ θλιβερή η ιστορία της Όπελ, ελπίζω να βρεθεί μια λύση, αλλά για να κλείσω θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι οι κατασκευαστές ακολουθούν τους πελάτες και όχι αντίστροφα. Και αυτό είναι ο σημαντικότερος λόγος για κάποιες ε, σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Αν ε, συρρυκνώνεται η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, ε, οπωσδήποτε και αυτό παίζει ρόλο. Και κάποιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετώπισαν κάποια δύσκολα προβλήματα. Τέλος, ε, μια ακόμη παρατήρηση σχετικά με το πεδίο αυτό έντασης που υπάρχει μεταξύ διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Μορέιρα έκανε την ερώτηση αυτή. Ο γύρος της Ντόχα από το 2009, εδώ και 9 χρόνια, ε, συνεχίζεται χωρίς να έχει ακόμη εξευρεθεί λύση. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, είμαι υπέρ των πολυμερών διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο ο γύρος της Ντόχα τα αναπτυξιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται εκεί θα πρέπει να διατηρηθούν και πιστεύω ότι σε ένα πολυμερές πλαίσιο ε, διασφαλίζεται και κάποια δικαιοσύνη για το διεθνές εμπόριο. Μέχρι να ε, ε, ολοκληρωθεί ο γύρος τέλος 2010-2011 ε, θα δούμε ε, τι θα ε, γίνει. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε και τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Όμως δεν πρέπει αυτές να ξεπεράσουν το πλαίσιο της Ντόχα. Οι αποφάσεις της Ντόχα δεν πρέπει να υπονομευθούν εννοώ. Και αυτό και εδώ μέσα εμπίπτει και η ΣΕΣ με την Νότιο Κορέα. Η, η πολυμερής διάσταση δεν υπονομεύεται ε, γιατί αν γινόταν αυτό θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις, πράγμα που δεν μπορεί να είναι σκοπός των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Μετά την παρέμβαση και του Επιτρόπου ολοκληρώνεται η συζήτηση. Μια και εξαντλήσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η επόμενη σύνοδος θα αρχίσει αύριο, 5η, 11 Φεβρουαρίου 2010, από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι τις 5. Μάλιστα, έχουμε το, το σχέδιο μερίσας διάταξης και στο έγγραφο και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.